Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Who came. Καλωσορίζω όλους εσάς που ήρθατε πουρνό-πουρνό ε, για την αρχή της συνεδρίασης. Ε, σημαντικότεροι είναι παρόντες, λέει ο κύριος Σαμαρζέ. Ναι, ναι, καλωσορίζουμε και όλους τους συναδέλφους ό,τι ώρα και να έρθουν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Λοιπόν, Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη για τη σημερινή συνεδρίαση. Μπορούμε να την εγκρίνουμε, παρακαλώ. Δεν βλέπω να διαφωνεί κανεί. Εγκρίνεται το σχέδιο τη ημερήσια διάταξη. Ω έχει. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Σχέδια πρακτικών τη 17η και τη 22η Ιανουαρίου. Διατίθενται ω συνήθω ηλεκτρονικά και προτείνω να θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Πρέπει να σας πω λίγα λόγια. Για το χθεσινό τριμερή διάλογο, χθες το βράδυ αρχίσαμε για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων Συναντηθήκαμε την Επίτροπο, την κυρία Κρέτσου, που εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τον Υπουργό Πλάμ από το Συμβούλιο. Ήταν from, from the Council. Και ήταν και πολυάριθμες και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις διαπραγματευτικές μας θέσεις. Εμείς λέω και εμείς και το Συμβούλιο εννοώ. Ακούσαμε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επί των θέσεων αυτών και στο τέλος της συνεδρίασης διαπραγματευτήκαμε το χρονοδιάγραμμα για τις τεχνικές συνεδριάσεις και τους πολιτικούς τριμερείς διαλόγους. Τι προγραμματίζουμε λοιπόν μέχρι τα μέσα Μαρτίου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, διότι μέσα Μαρτίου πρέπει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις λόγω των διαδικασιών στην Ολομέλεια τρεις ε, συνεδριάσεις πολιτικού τρίμερους διαλόγου θα έχουμε. Η πρώτη ήταν χτες, η επόμενη θα γίνει στις 22 του μηνός και η τρίτη στις 6 Μαρτίου. Και εκτός αυτών και μεταξύ των πολιτικών συνεδριάσεων θα έχουμε τουλάχιστον τρεις τεχνικές συνεδριάσεις για να δούμε μήπως έχουμε κάποιες θέσεις που να είναι τόσο κοντά ώστε να μπορούν να εγκριθούν κατά τη διάρκεια των τριμερών ε, πολιτικών διαλόγων. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής συνεδρίασης και αναμένουμε στις 25 του μηνός, όχι στις 22, να μας εξηγήσει το Συμβούλιο ποια θα είναι η τελική του αντίδραση και την αναμένουμε από πλευρά του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματά τους. Αυτό θα επηρεάσει άμεσα τη διαδικασία εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και στην Ολομέλεια για τον λόγο κανονισμό. Αυτά. Άλλη ανακοίνωση δεν έχω. Θα προχωρήσουμε τώρα στη μέση διάταξη. Το επόμενο σημείο είναι έκθεση για προϊόντα τα οποία δίνανται να τύχουν απαλλαγή σημείωση της εισφοράς θαλάσσης. Το 2014 ενέκρινε το Συμβούλιο μια ε, ε, πρόταση να επεκταθεί και να παραταθεί αυτή η ρύθμιση ε, μέχρι το 2020. Πρόκειται για προϊόντα που παράγονται σε κάποιες υπερπόντιες εκτίσεις και διαμερίσματα της Γαλλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης του Συμβουλίου, ε, το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2018 έκανε την πρότασή της για να τροποποιηθούν οι διατάξεις αυτές. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας τα εξηγήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. are indirect tax imposed on produced and imported into French outermost region Πρόκειται για προϊόντα ε, ε, Μαρτινίκας, Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όμως, ορισμένες αποκλήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές το Δεκέμβριο του 2004 όπου προβλέπεται πλήρης απαλλαγή ή μείωση του ύψους του συγκεκριμένου αυτού φόρου θαλάσσης. Έτσι, να, έτσι ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση με τα ίδια προϊόντα τα οποία παράγονται επί τόπου για να καλυφθεί η διαφορά η οποία οφείλεται στην ε, ε, μεγάλη απόσταση στην οποία βρίσκονται οι συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτά ε, γίνονται εφικτά με βάση το άρθρο 349. Προβλέπεται επίσης να ελέγχεται στο μέλλον η συγκεκριμένη δραστηριότητα και οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα που έχουν σαν στόχο να καλύψουν την υστέρηση των απομεμακρυσμένων περιοχών. Η Γαλλία ζήτησε να ανανεωθεί, να ενημερωθεί ο κατάλογος των προϊόντων που ε, καλύπτονται από τις εξαιρέσεις αυτές. προστίθενται 50 νέου τύπου προϊόντα έτσι ώστε να αλλάξει ο κατάλογος αυτός. Η Επιτροπή έχει επίσης προετοιμάσει μία έκθεση προς το Συμβούλιο The This proposal concern Προβλέπεται μια τεχνική προσαρμογή στο παράρτημα της απόφασης αυτής. Αυτό δεν επηρεάζει το περιεχόμενο ε, της ε, ρύθμισης αυτής, απλά αλλάζει τον κατάλογο, συμπληρώνει τον κατάλογο των προϊόντων τα οποία παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Η προσαρμογή αυτή είναι απαραίτητη γιατί τα τοπικά προϊόντα, αυτά που παράγονται τοπικά, εκτίθενται θα έλεγα σε ανταγωνισμό με εισαγόμενα προϊόντα, κάτι το οποίο δημιουργεί απειλές εις βάρος των τοπικών προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν η φορολογία στις απομεμακρυσμένες αυτές ε, πόνο, αυτόνομες περιοχές πρέπει να προστατευθούν διότι αλλιώς θα είναι καταστροφικές οι συνέπειες στις ε, επιχειρήσεις τις τοπικές. Έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για τους νέους. Προβλέπετε λοιπόν να υπάρξει και μία πλήρης συζήτηση εκ νέου της πρότασης αυτής όταν έρθει προς ανανέωση. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019. Έχουμε ξεκινήσει μια εξωτερική μελέτη, έχουμε ζητήσει να ολοκληρωθεί μια εξωτερική μελέτη, έτσι ώστε να μάθουμε αν το θέμα αυτό εξακολουθεί να έχει την σημασία την οποία προβλέπαμε. Η πρόταση αυτή έχει υποστηριχθεί από τις ομάδες εργασίας στις αυτόνομες αυτές περιοχές. Υπάρχουν και τρία λάθη σε επίπεδο ε, αριθμών. We thank you the, the committee for examining this, uh, this proposal. And uh, if you are δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Στις 17 Ιανουαρίου η συντονίστρια μας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την συντομευμένη, απλοποιημένη διαδικασία χωρίς τροπολογία, το 15-3. Και η πρόταση την οποία κάνω είναι να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροπολογίες. Η Σκιώδης πρώτα, ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Πονγκά ο οποίος όμως δεν είναι παρόν, αλλά έχει στείλει μία επιστολή λέγοντας ότι υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει λοιπόν με βάση το 15.1 χωρίς τροπολογίες την υιοθέτηση της πρότασης και ζητά να ψηφιστεί το ταχύτερο δυνατόν στην Ολομέλεια η πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Πογμπά. Ο κύριος ε, έχει το λόγο εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, εμείς υποστηρίζουμε την απλοποιημένη αυτή διαδικασία. Τον Ιούλιο του 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση που είχα προτείνει κατόπιν πρόταση τη Επιτροπή Ρέτζη για την εφαρμογή του άρθρου 349 που ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη, υπόψη της αυτό το άρθρο καλύτερα στο σύνολο νομοθετικών της προτάσεων. Επίσης η Επιτροπή μας το Σεπτέμβριο του 2018 οργάνωσε μια αποστολή στην Ρεϊνιόν και διαπίστωσε επί τόπου ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες ε, για τους παραγωγούς σε αυτές τις ε, πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Ε, οι νέες προτάσεις της Κομισιόν κατόπιν βεβαίων, βεβαίως ε, αρχικής πρότασης ενός κράτους μέλους της Γαλλίας πάνε προς την κατεύθυνση αυτή θα επιτρέψουν σε περισσότερα τοπικά προϊόντα, οπροκυπευτικά, έπιπλα ξύλινα να χρήζουν κάποιων εξαιρέσεων, κάποιων φοροαπαλλαγών σε αυτές τις περιοχές. Θα ενθαρρύνει αυτό την οικονομική δραστηριότητα, θα βοηθήσει τα τοπικά μας προϊόντα απέναντι σε έναν ανταγωνισμό ε, αυξανόμενο και που μπορεί να διακυβεύσει την ύπαρξη των τοπικών αυτών επιχειρήσεων ενώ ο παραγωγικό ιστός στις συγκεκριμένες περιοχές ε, είναι εξαιρετικά ισχνός και περιορισμένος. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν θα βοηθήσει την τοπική βιομηχανία να συνεχίσει να αναπτύσσεται ενώ ο κλάδος αυτός ε, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή δυσκολίες και βεβαίως όλα αυτά εγγράφονται σε ένα πλαίσιο ανεργίας, ε, σημαντικών ποστών ανεργίας, ιδιαίτερα για τους νέους από τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρώπης. Βεβαίως πολλά άλλα μέτρα χρειάζονται. Θα γίνει μια συζήτηση, όπως είπε και η Κομισιόν το 2019, για το μέλλον αυτού του καθεστώτος. Για την ώρα όμως, εμείς πρέπει να επικυρώσουμε αυτές τις εξαιρέσεις, τις παρεκκλήσεις που προτείνονται η ομάδα μας ε, πάντως ε, τις υποστηρίζει απολύτως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βάνσκου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει ο Μανσκούρ. Όπως και η προηγούμενη μητή θέλω να υπενθυμίσω τον πολύ κρίσιμο ρόλο του Κοινοβουλίου μας για να παραμένουν αγωνιστικές ε, αυτές οι επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και αυτό ε, έχει αντίκτυπο. Αυτό που μας προτείνεται σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα μεγαλύτερο εύρος εξαιρέσεων και, και μείωσης ε, της φορολόγησης που θα βοηθήσει ε, τις τοπικές επιχειρήσεις ε, και να αντιμετωπίσουμε έτσι και την ανεργία, ιδιαίτερα την ανεργία των νέων. Καλό τους συναδέλφους να φροντίσουν ή μπας περιπτώσει να μην αντιταχθούν σε αυτή την απλουστευμένη διαδικασία που μας προτείνεται έτσι ώστε στην Ολομέλεια γρήγορα να υπάρξει θετική γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Ο κύριος Ρόπε έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι αυτές οι περιοχές, αυτά τα νησιά χρειάζονται υποστήριξη. Αυτή είναι η γεωγραφική τους θέση. Ε, δεν φταίνε οι ίδιοι που μένουν εκεί. Έχουν μικρότερες δυνατότητες. Εκεί είναι περιορισμένη η ανταγωνιστικότητά τους Εάν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους παραγωγούς, τους τοπικούς παραγωγούς, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αρχές της πράσινης οικονομίας, ε, των μικρών κυκλωμάτων, μικρών αλυσίδων διανομής, καλό θα ήταν ε, να εφαρμοστούν αυτές οι εξαιρέσεις. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίδιοι για όλους. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν έχουν όλες οι χώρες τα ίδια χαρακτηριστικά, ούτε βεβαίω την ίδια γεωγραφική θέση. Εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πάρουμε και τις ε, κατάλληλες αποφάσεις γι' αυτό έγινε αναφορά στην ενεργεία των νέων. Και βεβαίως αυτό συνδέεται άμεσα και με την μετανάστευση για οικονομικούς λόγους. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα λύσουμε για να μένουν οι άνθρωποι σπίτι τους, να μην φεύγουν, να μην μεταναστεύουν, να αναπτύσσουν η οικονομία τους εκεί. Δεν μπορούν να ισχύουν λοιπόν οι ίδιες προϋποθέσεις παντού. Στις κάτω χώρες δεν είναι τα πράγματα όπως ε, αλλού, σε άλλες χώρες. Υπάρχουν διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να σκεφτεί κατά πόσο οι κανόνες και οι αρχές οι δικές μας αρκούν για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει σύγκληση και ε, ότι θα εξασφαλίσουμε τους ίδιες επίπεδο ανάπτυξη σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις εξαιρέσεις. Εάν αφήσουμε αυτές τις συγκεκριμένε ε, περιοχές την τύχη τους, εκεί θα, πάψει, θα πάψει να υπάρχει παραγωγή. Θα είναι απλώς εκεί όσοι δεν μπορούν να φύγουν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας και το ευρύτερο πλαίσιο. Οι χώρες της Βαλτικής, οι χώρες του Νότου, οι, χώρες, οι ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εξωτερικά σύνορα με τρίτες χώρες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Η γεωργία ποικίλει από χώρα σε χώρα. Οι άμεσες πληρωμές δεν είναι ίδιες. Κάποιοι αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους και πάνε αλλού για αυτό το λόγο. Και εκεί λοιπόν το να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες για όλους δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Οι χώρες που είναι στον πυρήνα της Ένωσης και οι χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια δεν μπορούν να ακολουθούν σίους κανόνες. Κάποιες χώρες είναι πιο απομακρυσμένες, έχουν εξωτερικά σύνορα, δεν μπορούν να αναπτύξουν τις ίδιες δραστηριότητε, δεν μπορούν και να ακολουθήσουν τους ίδιους κανόνες. εάν θέλουμε να περιορίσουμε και το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης, της οικονομικής αυτής εσωτερικής μετανάστευσης, νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μια νέα εποχή, την, την περίοδο 2021-2027, αυτή τη νέα περίοδο, την οποία θα αφιερώσουμε στο να επιλύσουμε το θέμα της σύγκλησης μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο δεν θα πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς τις περιφέρειες, ιδιαίτερα τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και να μειώσουμε και τη χρηματοδότηση και αυτό λάθος ε, θα ήταν. Ευχαριστώ. Υπάρχει υποστήριξη για την έκθεση της Κομισιόν και για την απλοποιημένη διαδικασία όμως είναι καθήκον μου να ρωτήσω για τελευταία φορά αν υπάρχουν αντιρρήσεις για να εγκριθεί αυτή η απλουστευμένη διαδικασία. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν αυτομάτως η έκθεση και θα ε, σταλεί στην Ολομέλεια και ελπίζουμε να ψηφιστεί εκεί το συντομότερο δυνατόν για να υποστηρίξουμε αυτές τις περιφέρειες διότι αυτό που θέλουμε είναι να υποστηρίξουμε την παραγωγικότητα τις δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση εδώ στην Επιτροπή Ρέτζη και προχωράμε. Λοιπόν, το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη είναι μια έκθεση δική μου και πάλι ως πρόεδρος έχω αυτή την ε, έκθεση, μπορεί για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Την 1η Φεβρουαρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια νέα πρόταση προς τροποποίηση ε, του τρέχοντος κανονισμού κοινών διατάξεων. Η τροποποίηση αυτή αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων για το 2019 για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μετά τις ε, συζητήσεις για τον προϋπολογισμό για το 2019. Θα ήθελα να δώσω λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σύντομη εξήγηση και παρουσίαση του θέματος και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ο κύριος Ντιπιέ Τραντόνιο και ελπίζω να το προφέρω σωστά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Καταρχάς, ε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, για την ταχεία ε, εξέταση και έγκριση αυτού του θέματος είναι σημαντικό και για μας και για όλη την Ευρώπη αλλά κυρίως για τα κράτη-μέλη εκείνα που εξακολουθούν να πλήττονται από την ανεργία των νέων. Πολύ σύντομα, η πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο, όπως είπατε, ε, αφορά και αντανακλά τη συμφωνία για την αύξηση του προϋπολογισμού για το ε, οικονομικό έτος 2019 είναι επιπλέον 116,7 εκατομμύρια ευρώ και προφανώς αυτό αντανακλάται και στο ειδικό κονδύλιο και στο κανονισμό ΣΥΠΙΑ για την τροποποίησή του. Το δεύτερο στοιχείο ανταποκρίνεται σε μια έκκληση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά διατάξεις που διευκολύνουν ε, επιπλέον ποσά και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 εδάφιο 5 του κανονισμού περί γενικών διατάξεων που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να μεταφέρουν μέχρι και το 50% ε, των κονδύλιων αυτών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Αυτά μπορεί να ακούγονται τεχνικά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ότι επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη και σε προγράμματα που τρέχουν να συνεχίσουν και να μην ε, αφαιρέσουν πόρους από μέτρα από που ήδη έχουν δεσμευθεί και να φροντίσουν μετά την αύξηση που ε, προώθησε το Κοινοβούλιο στη Συμφωνία του Προπολογισμού να συνδυάσουν τι δαπάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Σα ευχαριστούμε για την ταχεία διεκπαιρέωση και την ε, προστιμένη διαδικασία που επιλέγετε για να περάσει γρήγορα από την Ολομέλεια και εμεί φυσικά προσβλέπουμε στην έγκριση. Ευχαριστώ πολύ οι συντονιστές αποφάσισαν ακριβώς να προχωρήσουμε με απλουστευμένη διαδικασία και να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη τη σημερινή, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ταχεία διαδικασία, αλλά καταλαβαίνουμε τη σημασία και του θέματος και της ε, ταχείας αντίδρασης όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο σκιώδης ηγητής εξ ονόματος σοσιαλιστών και δημοκρατών, η συγκήτρια είναι η κυρία Κλέρ, και δηλώνει πλήρη υποστήριξη στην έκθεση αυτή και την απλουστευμένη διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχετε άλλα σχόλια. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μερικές συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απασχόληση των νεων Υπάρχουν ήδη κάποια κράτη-μέλη όπου δεν αρκεί να συζητάμε απλώ τη δημιουργία θέσεων απασχόληση ε, για τους νέους. Θέσεις εργασίας θέλουμε, αλλά και ποιοτικέ με καλές αμοιβέ, γιατί αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, υπάρχουν περιπτώσεις και καταστάσεις όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με μαζική ε, έξοδο των νέων και μετανάστευση για να ε, βρουν πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Το θέμα δεν είναι να βρεις μια δουλειά και ό,τι να είναι, αλλά να μπορείς να ζεις από τη δουλειά αυτή. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μέτρα. Να λάβουν μέτρα, Έτσι ώστε να μην υποχρεώνται οι νέοι να μεταναστεύουν για να βρουν δουλειά. Αν δεν μπορείς από το μισθό σου να πληρώνεις ε, ένα τραπεζικό δάνειο ή το νίκη σου ή να κάνεις διακοπές, τι να το κάνεις να δουλεύεις. Επίσης αντιμετωπίζουμε μια τεράστια κρίση σε σχέση με την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Αυτή είναι μια κατάσταση ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν δουλειές στη Γεωργία ε, και η κατάσταση είναι δραματική και θα πρέπει σε όλη την Ευρώπη να φροντίζουμε την απασχόληση των νέων. Η ανάπτυξη της ε, γεωργίας ε, με τον τρόπο που γίνεται δεν διευκολύνει προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, θέλω να το δούμε λίγο ε, πιο αναλυτικά και σε μεγαλύτερο βάθος αυτό το θέμα, ιδιαίτερα της ε, ανεργίας των νέων. Ζούμε σε ένα ενιαίο χώρο, τα περισσότερα κράτη είναι και κράτη-μέλη του Σέγγεν, άρα ελεύθερη κυκλοφορία είναι ε, απεριόριστη ακριβώς για ε, νέους που θέλουν να, ε, να ζητήσουν δουλειά σε άλλη χώρα από την πατρίδα τους. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Υπάρχει διαρροή εγκεφάλων και φεύγουν και καλά εκπαιδευμένοι και μορφωμένοι και υψηλή εκπαίδευση και ε, πολύ ειδικευμένοι εργαζόμενοι για να πάνε σε χώρε που πληρώνονται καλύτερα. Και στι φτωχέ χώρε λείπουν λοιπόν εργαζόμενοι με μεγάλη ειδίκευση στι νέε τεχνολογίε, στι ψηφιακέ τεχνολογίε. Ε, και αυτές οι χώρες που είναι σε καλύτερη μοίρα εξακολουθούν να αναπτύσσονται ενώ οι άλλες μένουν πίσω. Έχουν καλύτερη οικονομία, οι μεν πληρώνουν καλύτερους μισθούς και ε, προσελκύουν ε, και απορροφούν νέους ανθρώπους με πολύ καλή εκπαίδευση και κατάρτιση. Και χώρες περιφέρειες ε, πλήττονται. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει εδώ τις χώρες της Βαλτικής, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, χώρες οι οποίες αδειάζουν γιατί ε, ε, είναι τα κίνητρα πολύ καλύτερα σε άλλες χώρες. Φεύγοντας λοιπόν αυτός ο κόσμος, χειροτερεύει η κατάσταση στις χώρες. Είναι φαύλος κύκλος. Υπάρχουν και θέματα φοροαποφυγής και τα λοιπά. Υπάρχει μια εταιρεία που έχει την επίσημη έδρα της σε ένα κράτος, η παραγωγή βρίσκεται κάπου αλλού, τα κέρδη παράγονται επίσης κάπου αλλού και οι φόροι καταβάλλονται σε άλλη χώρα. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε, την επένδυση στους νέους. Και μια χώρα θα πρέπει να λαμβάνει ενισχύσεις Ε, και να αποζημιώνεται, γιατί μια χώρα έχει εκπαιδεύσει ένα νέο μηχανικό, ένα νέο γιατρό, ο οποίο σηκώνεται και φεύγει. Η χώρα έχει επενδύσει όμω επάνω του. Τι θα γίνει, έχει επενδύσει στην εκπαίδευση και στη μόρφωση των πολιτών. Θα πρέπει να αποζημιώνεται. Η ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να ε, είναι μια διαδικασία δούνε και λαβεί γιατί οι ε, πλούσιε χώρε απορροφούν όλο το δυναμικό ε, των ε, περιφερειακών κρατών όπου θα παραμείνουν μόνο συνταξιούχοι, ε, άνθρωποι με χαμηλή μόρφωση και χαμηλές δεξιότητες και προσόντα και δεν μπορεί να προχωρήσει μια περίπλοκη οικονομία. Άρα θα ενταθεί ακόμα περισσότερο αυτή η διαφορά, η φτώχεια και το χάσμα. Ξέρω ότι υπάρχει πολιτική συνοχή για να τα αντιμετωπίσει αυτά, αλλά δεν βοηθάει τη συγκεκριμένη κατάσταση για να ξεπεραστούν αυτές οι διαφορές που συσσωρεύονται. Γι' αυτό στο μέλλον ε, θα πρέπει να αλλάξουμε τακτική και να βρούμε άλλους τρόπους. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος? Ε, όχι. Λοιπόν, οφείλω επίσημα να ζητήσω αν υπάρχουν αντιρρήσεις στην πρόταση κανονισμού. Όχι. Η έκθεση λοιπόν αυτόματα θεωρείται δεκτή και παραπέμπεται στην Ολομέλεια. Ελπίζω το ταχύτερο δυνατόν να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη. Κατεξουσιοδότηση πράξη 481 του 14 δαπάνες για προγράμματα συνεργασίας. Θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την κατεξουσιοδότηση πράξη και μετά θα έχουμε μία συζήτηση μεταξύ των μελών και ίσως και κάποιες ερωτήσεις. Κυρία Βάγνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την κατεξουσιοδότηση πράξη. Είναι σχετικά τεχνική, οφείλω να ομολογήσω, η πρόταση αυτή. Ενθυμίστε την πρόταση, την πρόθεση, τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση Omnibus, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των δικαιούχων που ζητούσαν περαιτέρω απλοποίηση. Ήταν μια πολύ στοχευμένη διαδικασία απλοποίησης. Οι τροπολογίες τέθηκαν σε εφαρμογή στις 2 Αυγούστου. Αυτές οι τροποποιήσεις απαιτούν και αλλαγές σε επίπεδο δευτερογενούς νομοθετικής ε, ρύθμισης. Δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις, τις οποίες έχετε μπροστά σας σήμερα η δημιουργία μιας νέας τρίτης νομοθετικής πρότασης και μια εφαρμοστική πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή. Είναι ουσιαστικά επιμέρους ρυθμίσεις συνέπειες της αλλαγής τους κανόνες μέσω του Όμνιμπους. Και υπάρχουν και αρκετές διευκρινήσεις. Σχετικά με την συγκεκριμένη αυτή πράξη, τη σχετική με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών στα προγράμματα συνεργασίας. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δείτε και τα δύο αυτά στοιχεία συνδέονται με τις αλλαγές οι οποίες έχουν υπάρξει σε σχέση με τις απλοποιήσεις ε, ε, μέσω της αποφάσεως Omnibus. Προβλέπεται λοιπόν μία αναδιάρθρωση των άρθρων που στηρίζουν και αναφέρονται στην πράξη αυτή. Και δεύτερον, κάποιες αλλαγές που οφείλονται στη δυνατότητα πληρωμών με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η αναδιόρθρηση λοιπόν της απλοποιημένης ενιαίας μορφής πληρωμής απλοποιείται και οι αλλαγές που γίνονται έχουν σχέση με μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση part-time, επιμέρους απασχόληση, πώς υπολογίζεται. Γιατί πολλές φορές στις συμβάσεις απασχόλησης υπάρχουν κάποιες επιμέρους συμφωνίες Ο υπολογισμός των πληρωμών στο προσωπικό το οποίο απασχολείται προσωρινά γίνεται μέσω ε, της χρήσης των δικτών μέσου εισοδήματος όπως επίσης και της μέσης διάρκειας απασχόλησης μέχρι τώρα και το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Καλώς. Υπάρχει κάποιο σχόλιο λέει η Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν ε, θέματα. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει την δυνατότητα να θέσει εντηρήσεις. Η προθεσμία είναι η 7η Απριλίου. Μπορούμε να καθυστερήσουμε την πρόταση αυτή για ένα δίμηνο. Υπάρχουν μέλη τα οποία να διαφωνούν. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Έχει κλείσει λοιπόν η συζήτηση για την κατεξουσιοδότηση αυτή πράξη. Περνάμε με την επόμενη, στην οποία ήδη αναφερθήκατε άλλωστε. Τροποποίηση του 480, του κανονισμού 480. Αλλαγές στο CPR 2014-2020 μέσω της νομοθετικής ρύθμισης Omnibus. σε σχέση με την καταγραφή ε, δημοσίων πιστοτικών ιδρυμάτων, κρατικών επιδοτήσεων και ακροάσεων, ελέγχων λογιστικών. Για αυτήν την συγκεκριμένη κατεξουσιοδότηση πράξη, όπως και για την προηγούμενη, στην ουσία εφαρμόζουμε τις αλλαγές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί ήδη μέσω της πρότασης Omnibus. Είναι αρκετοί οι τομεί οι οποίοι καλύπτονται από την συγκεκριμένη αυτή κατεξουσιοδότηση πράξη. Είναι ουσιαστικά τεχνικές συνέπειες των προβλεπωμένων από το Omnibus. Οι νέες επιλογές οι εφαρμοστικές σε σχέση με την αλληλοεπίδραση και τον συνδυασμό του ΕΦΣΙ από τη μία και των διαφθορτικών ταμείων από την άλλη είναι κάτι το οποίο οργανώνεται και παρακολουθείται. Επίσης ε, τίθενται κανόνες σε σχέση με την διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των εσωτερικών ή εξωτερικών επενδυτών. Και το τρίτο στοιχείο αφορά την ε, δίκαιη μεταχείριση των διεθνών πιστοτικών ιδρυμάτων μέσω των διευκρινήσεων οι οποίες γίνονται στο βασικό άρθρο του CPR. Ένας άλλος τομέας στον οποίο προβλέπονται κάποιες τροποποιήσεις είναι η αντιμετώπιση των προγραμμάτων τα οποία είναι κερδοφόρα σε σχέση με ε, τις κρατικές επιδοτήσεις. Διευκρινίζεται λοιπόν εδώ ότι η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει ε, για περιπτώσεις όπου τα προγράμματα είναι καρπός κρατικών επιδοτήσεων. Επίσης, ε, μπορεί να γίνονται λογιστικοί έλεγχοι σε σχέση με τα προγράμματα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει πάντα το θέμα εδώ του ε, απλοποιημένου, των επιλογών πληρωμών των απλοποιημένων, λόγω ακριβώς αυτών των καταποκοπήν ποσών που προβλέπονται και στα πλαίσια της πρότασης ε, Omnibus. Ορισμένες ε, μορφές λογιστικού ελέγχου προβλέπονται επίσης. Προβλέπεται το πώς ακριβώς θα σχεδιαστεί ο λογιστικός έλεγχος όταν δεν εφαρμόζονται πλήρως οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές έτσι ώστε οι ενέργειες ή δράσεις να είναι ε, με σαφή ε, οικονομική ε, κάλυψη. Προτάσεις, γίνονται προτάσεις σε σχέση με την επιλογή των τμήματων, των δειγμάτων στα οποία θα γίνει έλεγχος και θα πρέπει οι επιλογές των δειγμάτων αυτών να αντικατοπτρίζουν αντικειμενικά τις αλλαγές που έχουν προβλεφθεί στο CPR. Και υπάρχουν επίσης και κάποιες προτάσεις αλλαγής στο παράρτημα 3 σε σχέση με το είδος του δικαιούχου και το είδος της χρηματοδότησης. Αυτά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι. Όχι. Πολύ ωραία. Να σας θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο βεβαίως μπορεί να φέρει αντίρρηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο πράξης κατοξιοδότηση. 12 Απριλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των αντιρρήσεων η οποία μπορεί να παρατεθεί ακόμα δύο μήνες. Έχει κάποιος αντίρρηση. Όχι. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις για αυτήν την πράξη, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ και προχωράμε στη μέρη διάταξη. Έχουμε τη χαρά να εξετάσουμε τώρα την μελέτη που ζητήθηκε από το τομέα Β, τομέα πολιτικής Β, ε, σε ό,τι αφορά την έρευνα στην, για την επιστροφή, Επιτροπή Ρέτζη, συγγνώμη, για το θέμα ψηφιακή ατζέντα και πολιτική συνοχής. Εμεί ε, ασχοληθήκαμε σε μεγάλο βαθμό με το πολιτισμικό πλαίσιο το τελευταίο διάστημα και έτσι αν αναγκαστήκαμε να συμπτύξουμε τι άλλε δραστηριότητέ μα. Δεν είχαμε ακούσει, παραδείγματο χάρη, τέτοιου είδου μελέτε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε κάτι σχετικό. Έχουμε και χρόνο για αυτή την παρουσίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να καλωσορίσω εδώ τη Ζουλή Πελεγκρά, η οποία είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Βιομηχανικών Μελετών στο Μιλάνο της Ιταλίας είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία η οποία κάνει μελέτες ό,τι αφορά σχέδια ε, δημόσιων επενδύσεων, ε, αξιολόγηση ε, σχέδιων υποδομών, υποστήριξη σε προγράμματα ανάπτυξης και πολιτικών κτλ. Θα ήταν καλό να μην περάσετε 20 λεπτά στην παρουσίαση σας, αν γίνεται. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει και η συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο στόχος της μελέτης που σας παρουσιάζω σήμερα το πρωί είναι να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια να παρουσιάσουμε μια κριτική ανάλυση της, πολιτική, της συμβολής της πολιτικής συνοχής και πιο συγκεκριμένα των διαθροτικών ταμείων στην ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη και στην ενιαία ψηφιακή αγορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Μας ζητήθηκε να εξετάσουμε και τις πρώτερες παρεμβάσεις των τομέα αυτών και βεβαίως να δούμε και την επόμενη προγραμματική περίοδο. Να πω δύο λόγια για τη μεθοδολογική προσέγγιση κατά τη μελέτη. Βασιζόμαστε σε μια εξέταση εγγράφων των πιο σημαντικών γράφων πολιτικής και αξιολογήσεων, μια ανάλυση των διαφόρων ε, μορφών ε, δαπανών, πέντε παραδείγματα ε, project επενδύσεων στο στην ψηφιακό τομέα και που χρηματοδοτούνται από την ΕΣΥΦ και μια σειρά από συνεντεύξεις κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσίασή μου ακολουθεί μια χρονολογική σειρά. Θα εξετάσουμε τις πρώτερες ε, παρεμβάσεις, θα εξετάσουμε ε, επίσης το τι συνέβη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος, και θα μιλήσουμε και για το μέλλον βεβαίως, τι θα συμβεί δηλαδή μετά το 2020. Θα ξεκινήσω τονίζοντας το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι προπομπός ε, σε ό,τι αφορά, είναι πρωτοπόρος ε, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια ε, συνοχής, δηλαδή πιο μακρισμένες περιοχές να μπορούν να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στην δεκαετία του 80 ήδη είχαμε τις πρώτες πρωτοβουλίες ε, και στην δεκαετία του 90, το 2000 ε, εμφανίστηκαν οι πρώτες στρατηγικές ψηφιακής πολιτική και τελικά είχαμε την έγκριση της ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη το 2010 και την ενιαία ψηφιακή αγορά το 2015. Από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ακολουθεί μια εξαιρετικά σταθερή προσέγγιση, έχει μια σφαιρική ε, εικόνα, δίνουμε έμφαση και στην παροχή ε, νέων τεχνολογιών, τις υποδομές αλλά και τη ζήτηση ψηφιακών τεχνολογιών από τους πολίτες, από τις επιχειρήσεις, από τις διοικήσεις, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, τις ψηφιακές κτλ. Μια σφαιρική προσέγγιση δημιουργεί έναν θετικό κύκλο όπου ε, η προσφορά ε, μεγαλώνει τη ζήτηση και τούμπαλιν. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό εδώ το θέμα της συμπερίληψης όλων στη διαδικασία αυτή. Τώρα, η εκτιμόμενη συνεισφορά του ΕΣΥΦ ε, είναι υψηλή. Ε, είναι πολλά τα κονδύλια που διατίθενται και βεβαίως ε, το περιφερειακό επίπεδο είναι το κατάλληλο για να μπορέσει να ακολουθεί μια σφαιρική προσέγγιση. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα η υποστήριξη της πολιτικής συνοχής ε, αυξήθηκε με τον καιρό από τα 1,2 δις στη δεκαετία του 90 στα 21,4 δις πλέον στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Να πω κάτι επί της μεθοδολογίας. Πρέπει να καταστήσω σαφές ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ε, όταν προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τις επενδύσεις ε, στον ψηφιακό τομέα και σε στατικό επίπεδο και σε δυναμικό επίπεδο, διότι έχει έναν οριζόντιο χαρακτήρα αυτή η επένδυση, εγγράφονται δηλαδή εντός άλλων επενδύσεων, είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να συνδυάσει κανείς, αλλάζουν ε, τα συστήματα αλλάζουν και, τα, και, η, ταξι, αλλάζει και η ταξινόμηση κατά τη διάρκεια τη κάθε προγραμματική περίοδου. Τώρα για την περίοδο 2000-2006 βλέπουμε ότι δόθηκε προτεραιότητα στις υποδομές. Ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν στη δεύτερη θέση. Για την περίοδο 2007-2013 Εδώ η προτεραιότητα δόθηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στις ε, εφαρμογές για τους πολίτες. Τώρα για την τρέχουσα περίοδο δώσαμε έμφαση και πάλι στις υποδομές και στη συνέχεια ηλεκτρονική δικυβέρνηση, ψηφιακές δεξιότητες. Μπορείτε όλα αυτά να τα δείτε σαφέστερα στη σελίδα 17 της έκθεσης. Με δύο λόγια τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής. Οι επενδύσεις του ΕΣΥΦ στις υποδομές νέων τεχνολογιών είναι ε, βασικός παράγοντας παρέμβασης στο συγκεκριμένο κλάδο. Είχαμε μια πρόσφατη αύξηση μάλιστα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Όμως, εάν δούμε μαζί τις επενδύσεις ε, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στα ψηφιακά, ψηφιακές δεξιότητες και στην ηλεκτρονική συμπερίληψη, ένταξη, είναι ένα, έχουμε ένα σταθερό έτσι, κομμάτι, μερίδιο των, των συνολικών ψηφιακών επενδύσεων. Περίπου 40% επίσης έξυπνες πόλεις, έξυπνα δίκτυα που αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και μην ξεχνάμε και την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι όμως χαμηλό αυτό το ποσοστό, αυτό το μερίδιο κατά τη διάρκεια της πραγματικής περίοδου. Να πω δύο λόγια και για τις γεωγραφικές ε, γεωγραφική κατανομή αν θέλετε μπορεί και πάλι στη σελίδα 78 εδώ να δείτε καλύτερα τα στοιχεία αυτά στην έκθεση βλέπουμε ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης ε, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση ε, στην ε, ψηφιακή τεχνολογία, ιδιαίτερα στην Ισπανία ε, τώρα κατά κεφαλήν η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι μπροστά. Ε, να δώσω κάποια στοιχεία. σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές οι δαπάνες για επενδύσεις ΕΣΥΦ είναι 113 κατά κεφαλήν 113 ε, ευρώ ανά άτομο δηλαδή 49 ευρώ στις περιοχές μετάβασης και 37 ευρώ στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Ποιες είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται όμως επί, επί που πέρα από αυτά τα συνολικά στοιχεία που σας παρουσίασα. Σε ποιο πλαίσιο λαμβάνουν χώρα αυτές οι περιφερειακές ψηφιακές επενδύσεις. Όπως γνωρίζετε είχαμε σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της, του ΕΣΥΦ και αυτό έχει επιπτώσεις για τις ψηφιακές επενδύσεις. Γίνεται μια προσπάθεια να έχουμε θεματικές συγκεντρώσεις, να υπάρχουν δηλαδή κάποιοι θεματικοί στόχοι και ένας από αυτούς σχετίζεται με τις ψηφιακές ε, επενδύσεις, είναι θεματική δύο. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις εξάντε αντέ, που έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές επενδύσεις. Ε, ε, ένας κοινό ε, κανονισμός ε, διευκολύνει τη χρήση των ταμείων και των διαφορών μέσων που έχουν, που έχουν θεσπιστεί για να έχουμε μια προσέγγιση που να βασίζεται ε, στους τόπους, στους διάφορους τόπους. Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση συνδυασμένα στοιχεία έχουμε εντοπίσει δύο βασικούς παράγοντες επιτυχίας πρώτο έχει να κάνει με τη σημασία του στρατηγικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τι ψηφιακέ επενδύσει. Αυτό μα επιτρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση που καλύπτει τι διάφορε διαστάσει τη σφαιρική προσέγγιση και περιλαμβάνει, μα δίνει δυνατότητα να συνδυάσουμε μια σειρά από στοιχεία, ευρυζωνικά δεξιότητε, ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το θετικό κύκλο στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Το δεύτερο, το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την ανάπτυξη συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, των διαφόρων ε, τεχνολογιών. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε τις κατάλληλες, τις απαραίτητες επενδύσεις, να καλύψουμε τις ε, ελλείψεις ό,τι αφορά τις διοικητικές δυνατότητες ή δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο η ανάλυση μας δείχνει ότι η διαδικασία θέσπισης ε, ε, υγιών ε, εταιρικών σχέσεων που οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι μια μακρά διαδικασία και δύσκολη. Πρέπει να, αυτό να, να το να διοικείται εκ των έσω και όχι εκ των απ' έξω. Τα παραδείγματά μας δείχνουν ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης δίνουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν και οι δύο αυτές προϋποθέσεις επιτυχίας. Πρέπει να υπάρξει μια η κατάλληλη στρατηγική προσέγγιση και να προωθηθούν ε, οι συμπράξεις αυτές και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να συνδυάσουμε και διάφορες μορφές χρηματοδότησης για να συμβεί αυτό. Να σας πω ακόμα μερικά ευρήματα. Έχουμε εντοπίσει κάποιους τομείς όπου η πολιτική συνοχή θα μπορούσε να προωθήσει καλύτερα την διάδοση της, ψηφιακή της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και σε τομές όπου κάποιες εφαρμόγες ε, νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες. Για το ERDF, το, το Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης, επικεντρώνεται κυρίως ε, στις ε, υποδομές νέων τεχνολογιών. Επίσης εντοπίσαμε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συμπληρωματικότητα μεταξύ ΕΖΙΦ και συνεργειών μεταξύ ΕΖΙΦ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Θα είμαι σύντομη σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων ε, ταμείων ε, και μεταξύ των διαφόρων ε, υποταμείων του ΕΖΙΦ, μια και αυτό δεν αφορά τόσο τον τομέα των νέων τεχνολογιών. Θα ήθελα απλώ να επιμείνω λίγο στο θέμα τη συνέργεια μεταξύ ΕΣΥΦ και του ορίζοντα 2020 μια συνέργεια η οποία δεν είναι τόσο προφανής πάντα θα υπάρξει όμως περαιτέρω εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι φτάνουμε στα συμπεράσματα σιγά σιγά. Η μελέτη μας Έρχεται ε, να επικυρώσει την, ε, στο σωστή προσέγγιση του συστήματος αυτού. Είναι προσαρμοσμένο για μια σφαιρική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές επενδύσεις. Η πολιτική συνοχή όμως πρέπει να επικεντρωθεί εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Υποστήριξη ε, των κατάλληλων στρατηγικών σε περιφερειακό επίπεδο για ψηφιακά ζητήματα και την σωστή σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο και πέρα από αυτό. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη υποστήριξη των σχεδίων επενδύσεων και τη υποστήριξη των πολιτι... τη άσκηση πολιτική και των διοικητικών δυνατοτήτων. Και το δεύτερο δεν πρέπει να ε, αναπτυχθεί, διωγγωθεί υπερβολικά σε σχέση με το πρώτο. Επίσης, στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ε, είναι ένα προνομιακό, ένας προνομιακός τομέας για να μπορέσουν, να μπορέσει να στεφθεί από επιτυχία το εγχείρημα, γιατί εκεί μπορεί να, να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση με συνέργειες, με συμπράξεις, ε, η οποία φέρνει αποτελέσματα. Επ' αυτής της βάσης εμείς έχουμε προετοιμάσει μια σειρά από συστάσει, Εδώ βλέπετε μια, κάποιες από αυτές, εν πάση περιπτώσει. Πρώτα απ' όλα μας φάνηκε απαραίτητο να ευθυγραμμίσουμε τα συστήματα διακυβέρνησης ε, και αποτελεσμάτων. Ε, για να συμβεί αυτό, καλό θα είναι να υπάρχει ένα έγγραφο πολιτικής που να αναφέρεται στους στόχους της στρατηγικής σε σχέση με την ψηφιακή ατζέντα και αυτά να μεταφράζονται σε συγκεκριμένου επιχειρησιακού στόχου. Ε, αυτό το έγγραφο θα προβλέπει και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του και των ευθυνών. Φαίνεται να είναι απαραίτητο επίσης να επανεξετάσουμε και το σύστημα της, ε, των προποθέσεων ex ante εκ των προτέρων θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την έξυπνη εξειδίκευση και σχετικέ στρατηγικέ, παραδείγματο χάρη, να πούμε ότι πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά εκεί στις ψηφιακέ επενδύσεις θα μπορούσε να είναι άλλη μια προϋπόθεση εξάντε αυτή μια άλλη προϋπόθεση θα μπορούσε να είναι αυτή που υπάρχει και τώρα ε, που έχει σχέση με τις υποδομές των τεχνολογιών που είναι περίπλοκες ε, και χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Φαίνεται επίση αναγκαίο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ ΕΖΙΦ και ΟΖΙ 2020 και βεβαίως η έξυπνη εξειδίκευση και σχετικές στρατηγικές ε, και εδώ φαίνεται να είναι το κατάλληλο εργαλείο για να συμβεί αυτό. μπορεί να γίνουν και βελτιώσει σε ρυθμιστικό επίπεδο για να υπάρξει σαφές ο διαχωρισμό μεταξύ ERDF και του Ταμείου ε, για την Περιφερειακή Ανάπτυξη που σχετίζεται με ψηφιακή στην ψηφιακή τεχνολογία στην Ήπεθρο. Θεωρούμε ότι η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών πρέπει να ε, διαδοθεί, να ενισχυθεί συγγνώμη, στον τομέα της οικονομίας της υπαίθρου αλλά και στην τομέα της κλιματικής αλλαγής τα έλεγα και νωρίτερα αυτά ε, μέσω συγκεκριμένων εστιασμένων προγραμμάτων και τέλος υπάρχει η ανάγκη να βελτιωθεί η βάση των γνώσεων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας ε, τα συστήματα παρακολούθησης πρέπει να βελτιωθούν να υπάρχουν περισσότεροι δείκτες που σχετίζονται με ψηφιακή απόδοση και τις δαπάνες βεβαίως. Οι δαπάνες με ψηφιακό ε, περιεχόμενο θα πρέπει να ε, σημειώνονται για να δείξουμε τον οριζόντιο χαρακτήρα ε, των ψηφιακών τεχνολογιών και σχετικών επενδύσεων. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο ερωτήσεις. Ο κύριος Όλμπρεχτ. Μια τεχνική ερώτηση έχω. Παρατηρώντας την πρόταση για τις νέες προτεραιότητες του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, διαπιστώνουμε ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι η πρώτη αλλά σε σχέση με τις επικοινωνίες και την μεταφορά και τις μεταφορές ψηφιοποίηση των συγκοινωνιών, των δρόμων, των αυτοκινοδρόμων, των σιδηροδρόμων. Περίεργο μου φαίνεται γιατί ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία της πληροφορίας, με την ψηφιοποίηση, με τον εξυγχρονισμό, είναι πρώτο. Τώρα γιατί το έχει βάλει ε, στις μεταφορές με τους δρόμους και τους σιδηροδρόμους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στο κεφάλαιο με τα ψηφιακά. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εμπειρογνώμονα για την παρουσίαση. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω την ανάγκη ανάπτυξης ε, της ψηφιοποίησης, ιδιαίτερα στις περιοχές της Υπέθρου. Είναι η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο πράγμα που ζητούν οι νέοι για να εγκατασταθούν στην Υπέθρο. Να έχουν πρόσβαση σε ένα γρήγορο ίντερνετ, σε ένα ευρυζωνικό. Αλλιώς δεν πρόκειται να εγκατασταθούν ποτέ οι νέοι ε, στην Ήπεθρο. Την περασμένη χρόνια, πέρσι, είχα πάει στην Ιρλανδία και δεν ήταν πάρα πολύ καλή η σύνδεση στο διαδικτύο ούτε στις πόλεις ούτε στην Ήπεθρο. Και θέλω να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες γιατί τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν τα κονδύλια που υπάρχουν έτσι ώστε να ε, διευρύνουν το δίκτυο του διαδικτύου και μάλιστα του ευρυζωνικού. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Επίση, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει γιατί δεν υποστηρίζονται παρκώ για να προωθούν την ψηφιοποίηση. Προηγουμένως μιλήσαμε για έλλειψη εργατικού δυναμικού. Γιατί λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Ευτυχώς στη Ρουμανία έχουμε πολύ καλό διαδίκτυο και πάρα πολύ καλή σύνδεση. Ε, μετά όμως συζητάμε τελικά ε, για τις ανάγκες όλης της Ευρώπης. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση για την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη και γενικά. Όλο και περισσότερα κονδύλια βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζουν ε, την ψηφιοποίηση. Και ακριβώς αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε επίσης ότι υπάρχει τεράστια διαφορά στην κάλυψη ανάλογα με ε, τη χώρα. Κυρίως για το γρήγορο διαδίκτυο και αναφέρθηκε και ο κύριος Μπούντα στη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις πόλεις και την Ήπεθρο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάλυψη στις πόλεις διαδικτυακή σε ποσοστό που φτάνει πλέον το 90%. Στην Ήπεθρο είναι περίπου το μισό. Πρέπει να κλείσει αυτό το χάσμα ανάμεσα στην Ήπεθρο και στις πόλεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ. Και βλέπω μια μικρή αύξηση, 5 με 10% στην ε, ατζέντα για την Ήπεθρο και το 70,5% έχει δεσμευθεί για τις έξυπνες πόλεις και τα έξυπνα χωριά που είναι η νέα πρωτοβουλία. Τι σημαίνει αυτό. Ότι βλέπουμε την Ήπεθρο συνολικά, σφαιρικά και θέλουμε να έχουμε τις βασικές υποδομές παντού, βασικές δεξιότητες παντού και μείωση της αστιφιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη και η παρουσίασή σας τώρα έδειξαν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα διάφορα ταμεία. Δεν, ξέρω γιατί κάνετε αυτή τη διάκριση ε, πόλεων και περιοχών της Υπέθρου Δεν είναι μόνο έξυπνες πόλεις, είναι και τα έξυπνα χωριά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως έννοια διάφορες μικρομεσαίες εταιρείε για να εγκαθίστανται εκεί με συνέργειες. Στην Ήπεθρο αυτό που χρειάζεται είναι δημόσιες επενδύσεις, ακριβώς για να δημιουργηθούν οι βασικές υποδομές που είναι προϋπόθεση για να επιτυχθούν όλες οι υπόλοιπε δραστηριότητες που χρειάζονται ε, ε, για να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού όπως είναι η ηλεκτρονική διοίκηση, διακυβέρνηση κλπ. Ε, τι έχετε λοιπόν στο μυαλό σας όταν μιλάτε για καλύτερη ευθυγράμμιση ή συνδυασμό ε, του Γεωργικού Ταμείου και του Ταμείου για την Ανάπτυξη Πέθρου. Ευχαριστώ. Ερωτήσει σχόλια, ο κύριος Ομαγζέ. Ευχαριστώ. Αυτό που ισχύει για τις περιοχές της Υπέθρου Ισχύει και για τις ιδιαίτερα απόμακρες περιοχές. Η ψηφιοποίηση είναι βασικό χαρακτηριστικό για τον απεγκλωβισμό των περιοχών αυτών, των νησιωτικών ιδιαίτερα. Βλέπω πολλά θετικά εδώ. Στην 34 σελίδα βλέπω ότι υπάρχουν ε, και κάποιες αντεδείξεις σε σχέση με αυτά τα οποία λένε οι υπερπότιες περιοχές. Η ηγεσία των υπερπόντιων γαλλικών περιοχών μας λέγουν ότι είμαστε στην κορυφή, ενώ ε, τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι έχουμε μεγάλο βαθμό ιστέρησης ε, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο πράγματι θα μας βοηθήσει. Ο κύριος Ρόπες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν την ε, την εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίασή της, διαπιστώνουμε ότι ο ψηφιακός τομέας πράγματι επηρεάζει με πολύ σημαντικό τρόπο στα θέματα της συνοχής. Στην παρουσίασή σας σχολιάσατε ήδη κάποιες πλευρές οι οποίες με οδήγησαν να σκεφτώ κάποια ε, από τα θέματα αυτά ε, πολύ περισσότερο. Η προσωπική μου εμπειρία ε, λέγει ότι όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα των περιφερειών τους, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Σαν παράδειγμα στο πρόγραμμα ηλεκτρονική υγεία, γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να δημιουργήσει κανείς ένα ιδανικό σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να υπάρξει ανταλλαγή χρηστών πρακτικών και εμπειριών ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό τα οποία έχουν συγκεντρώσει ε, περισσότερες εμπειρίες, που έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο, μπορούν να βοηθήσουν τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό είναι σημαντικό σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα όμως στον ψηφιακό τομέα. η ηλεκτρονική μας ατζέντα μερικές φορές επιτρέπει την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών και επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό ακριβώς η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι μια πρακτική η οποία θα έλεγα είναι ιδιαίτερα θετική. Αναφερθήκατε επίσης και στο θέμα της διαχείρισης των επενδύσεων και εδώ θα ήθελα ίσως κάποια περισσότερο σχόλια γύρω από το σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως να έχετε εντοπίσει κάποια προβλήματα τα οποία τίθενται. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί εκεί όπου τα προβλήματα είναι πιο σοβαρά. Σχετικά με την γεωργία πάρα πολύ συχνά λέγουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στον γεωργικό τομέα και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στις, ε, στις τεχνολογίες της πληροφορικής. Αλλά όμως βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να το κάνουν. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν και να γίνουν αποδοτικές. Να μην ξεχνάμε όμως ότι οι επιχειρήσεις αυτές αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι να παράγουν γεωργικά προϊόντα με ανταγωνιστικές τιμές. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος, αυτή είναι η βασική τους αποστολή. Σχετικά με τα μέσα και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν, αυτά εξαρτώνται από την συγκεκριμένη εταιρεία. Τι παράγει η εταιρεία, παράγει τράκτορες, παρά, ε, παράγει αγροτικά τρακτέρ, εν πάση περιπτώσει παράγει ε, ηλεκτρονικά προϊόντα, εξαρτάται από τη φύση της επιχείρησης. Εμείς απλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες δυσκολίες σχετικά ε, με την προμήθεια γεωργικών προϊόντων. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισόδημα των γεωργών αντιπροσωπεύει ε, το 50% του συνόλου του τομέα. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν για την βιομηχανία μας να λύσει κάποια από αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να μειωθούν ε, κυρίως ε, οι επιβαρύνσεις οι οποίες υπάρχουν εις βάρος των γεωργών. Και δεν θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να είναι υπεύθυνες έτσι ώστε να αγοράσουν τις πιο ακριβές και αποδοτικές τεχνολογίες. αλλά θα πρέπει η βιομηχανία να κάνει συγκεκριμένες καινοτόμες προτάσεις και να λύσει τα προβλήματά της. Πρέπει λοιπόν ε, οι υπεύθυνοι για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενωμένοι να παραγγέλνουν τα σωστά υλικά, τους σωστούς εξοπλισμούς και να εκμεταλλεύονται σωστά. Αυτό όμως δεν φτάνει. Νομίζω ότι η βιομηχανία στην Ευρώπη θα πρέπει και αυτή με τη σειρά της να λειτουργήσει πιο θετικά για τους γεωργούς. Υπάρχουν ταμεία κοινοτικά για την έρευνα, υπάρχουν ταμεία κοινοτικά για την καινοτομία και όλα αυτά τα ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το σημαντικό πρόβλημα που είναι τα εισοδήματα των γεωργών. Αυτά θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της γεωργίας μας. Αν κάποια από τα χρήματα αυτά τα στρέφουμε στην ψηφιοποίηση, τότε στο μέλλον μπορεί να αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Νομίζω ότι από αυτό θα ωφεληθεί και η γεωργία και η έρευνα και οι βιομηχανίες. Ερωτήσεις. Άλλη. Η κυρία Πελεγκρά έχει την ευκαιρία, έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε σε όλα τα σχόλια, τις προτάσεις και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Για ποιο λόγο η ψηφιοποίηση λέτε έχει μπει στις μεταφορές και δεν σας αρέσει. Εγώ ε, ε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε τις πρόσφατες εξελίξεις. Αυτό είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαι ε, η καλύτερη για να σας απαντήσω εγώ. Αλλά εκπλήσουμε κι εγώ όπως κι εσείς. Το λεπτό και ευαίσθητο θέμα της ψηφιοποίησης στην Ήπεθρο. Άκουσα διάφορα σχόλια γι' αυτό Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν είναι απολύτως ικανοποιητική. έως ε, προς την ψηφιοποίηση της υπαίθρου. Αυτό εν μέρη μόνο εξηγείται από τα ασαφή όρια των ταμείων, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου για την Ανάπτυξη της Υπέθρου. Δηλαδή για το ποιο είναι αρμόδιος για να χρηματοδοτήσει τι. Την ευρυζωνικότητα και τις υποδομές πληροφορικής και τεχνολογίας των κοινωνιών. Ε, και ότι αυτή η ασάφεια έχει καθυστερήσει τις ε, επενδύσεις. Αυτό εξηγείται εν μέρη μόνο από τα ταμεία. Αλλά οι επενδύσεις αυτές περιορίζονται στις υποδομές και δεν αφορούν μια καθολική, ολιστική, σφαιρική προσέγγιση. Γιατί δεν γίνεται, ε, καλά, δεν, δεν δίνεται απαραίτητη προσοχή στις δεξιότητες, τα ε, προσόντα που απαιτούνται, στο κατά πόσο είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτές να εκπαιδεύσουν ε, στα νέα επαγγέλματα και στις νέες δεξιότητες. Λοιπόν, για ποιο λόγο χρειάζεται να υπάρξει αυτός ο σαφής διαχωρισμός, γιατί πρέπει να ξέρουμε ο καθένας τι ευθύνε έχει και ποιος κάνει τι. Αυτό δεν αποκλείει όμως την ανάπτυξη ε, συνεργειών και συνεργασιών. Στην αρχή χρειάζεται ένα σαφής επιμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών και μετά να υπάρχει ένας μηχανισμό για συντονισμό μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Αφήνω για να τελειώσω τα θέματα της υπαίθρου από το Ότι δεν θα πρέπει να επενδύουν οι αγρότες στις ψηφιακές τεχνολογίες. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και το σημειώνω. Αλλά πώς να το πω. Το θέμα είναι να κάνουμε τη ζήτηση να συναντήσει την προσφορά ε, τεχνολογιών τέτοιων ψηφιακών. Υπάρχει ο κλάδος ε, για να παρέχει τις λύσεις, αλλά χρειάζεται και μια απόκριση ε, και ε, συνεργασία με τους αγρότες που θα ενημερώσουν τους αρμόδιους για τις πραγματικές τους ανάγκες. Εξού και η εταιρική σχέση που πρέπει να προωθεί για να είναι αποτελεσματικές επενδύσεις και στην Ήπεθρο. Επίσης, έγινε μια ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκφράστηκε κάποια απογοήτευση για τις προσπάθειες ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνώ. Μια πιθανή απάντηση εξήγηση θα ήταν η εξή. Η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλύπτεται από άλλα κονδύλια, από τα ταμεία. Από το σχέδιο Juncker ή το πρόγραμμα COSME. that's a hypothesis υποθέτω. Αλλά είναι ένα αποτέλεσμα της μελέτης που μας προξενεί εντύπωση. Νομίζω ότι απάντησα στις διάφορες ερωτήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ και για τα αντίγραφα της μελέτης που μας στείλατε. Έχουμε όλη τη μελέτη σε δύο μέρη και εάν υπάρξουν άλλα σχόλια και ερωτήσεις βεβαίως ε, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με την ημερησία διάταξη και περνάμε στο επόμενο σημείο, έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Έχετε λάβει ένα mail με τις αποφάσεις των συντονιστών που πάρθηκαν στη συνεδρία στις 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο μπορούμε να εγκρίνουμε αυτές τις αποφάσεις. Πολύ ωραία. Τώρα υπάρχει κάτι από τα διάφορα και ο κ. Βανίστελ Ρόι δεν είναι εδώ, δεν έχουμε και διάφορα. Μας λείπει, ναι, μας λείπει στο σημείο αυτό να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 21 ε, Μαρτίου, 5η, ακυρώσαμε τη συνεδρία στις 7 Μαρτίου, 21 Μαρτίου, λοιπόν 5η, 21 Μαρτίου το πρωί, 9 με 10 και μισή, με 12 και μισή. Αυτή ήταν η τελευταία πληροφορία για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους και καλή σας μέρα. Ολοκληρώνουμε.